Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, λοιπόν, να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσης διάταξης, δεν βλέπω αντιρρήσεις, ωραία. Ωραία. Πρόταση για μια ευρωπαϊκή σύνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Η Μαρή Χριστίνα Νοτού είναι η συγγήτρια και περνάμε στην ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Για να δούμε αν έχουν όλε οι ομάδε ε, την αριθμητική δύναμη που του αναλογεί. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, ακόμη. Α, είναι χαλασμένο. Καλά. Ωραία. Άρχεται και πάλι η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία πέρας. Ωραία, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 12. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ποιος, ποιος παρακαλώ. Θα πρέπει να μας πείτε πριν από την ψηφοφορία τι προτίθεστε να ψηφίσετε. Με το με δείχτε, δείχτε μας με χειρονομία. Πέρασε. 19 υπέρ 21 κατά 4 αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16. Α, 16, α, καταπίπτει. 17 υπέρ. Α, και η 17. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3. Καταπίπτει 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, όχι. Όχι, να ελέγξουμε τη 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εσείς, μάλιστα, σημειώνω. 23 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος. Η τέσσερα καταπίπτει. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22. Α, 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πριν ψηφίσουμε για την συνολική γνωμοδότηση, όπως λέει ο κανόνας εάν οι τροπολογίες των, των γνωμοδοτουσών επιτροπών ε, περιέχουν τροπολογίες τότε πρέπει να υπάρξει σύντομη ιτολόγηση επειδή δεν έχει εγκριθεί καμία τροπολογία δεν μπορεί να γίνει και καμία γνωμοδότηση οπότε δεν χρειάζεται καμία τελική ψηφοφορία οπότε θα στείλω αυτή τη γνωμοδότηση οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τελική ψηφοφορία και έτσι αποφασίσαμε του θέματος αυτού. Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τροπολογία το σύνολο των τροπολογιών απορρίφθηκε. Όμως, Υπάρχει μία τροπολογία του ΕΛΚ η οποία εγκρίθηκε, αν κατάλαβα καλά, με μία ψήφο διαφορά 23 υπέρ, 21 κατά, όχι, όχι λάθος έκανα, λάθος, εντάξει, συγγνώμη, ξεχάστε το αυτό που είπα. Πρόεδρος, έγινε δεκτή η απόσυρση της τροπολογίας, γι' αυτό δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία. Λίγη τη συνεδρία. Ευχαριστούμε πολύ.